στις 5 ε, Μαΐου με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατό του. Έγινε Ευρωβουλευτής το 2014, ήταν μέλος στην Επιτροπή Αναπτύξεως, στην Αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Αφγανιστάν. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω θερμότατα συλληπιτήρια όλων μας στην οικογένεια και τους οικείους του κ. Χανσιάντσεν.